Αγαπητοί και συνάδελφοι, ξαναπαίρνουμε τη σκητάλη εκεί που την είχαμε αφήσει χθε το βράδυ. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λιάντ Νιθιαντά για την κινητοποίηση του Ταμείου Προσαρμογή στην κινητοποίηση, στην, συγγνώμη, στην Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι πολύπλοκο το θέμα αυτό. Σχετίζεται με, την, ε, με, με το σούπερ μάρκετ της Λάρισας. Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν αυτή την αίτηση για χρηματοδοτική βοήθεια από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης στις 26 Νοεμβρίου 2015. Η αξιολόγηση περατώθηκε στις 14 Απριλίου 2016 από την Κομισιόν. Έγινε με ταχύ ρυθμό λοιπόν Ξέρουμε βέβαια τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχει η ελληνική οικονομία ήδη για 8 χρόνια και δεν έχει βγει ακόμα. Έχει μειωθεί σημαντικά και η κατανάλωση, έχει αυξηθεί στα ύψη η ανεργία. Το είδαμε και εμείς και το γνωρίζουμε και από γνωστούς μας ότι υπάρχουν ελλείψεις τροφίμων, ότι υπάρχουν προβλήματα με τους εργαζομένους. Επομένως δεν είναι καθόλου εκπληκτικό ότι αυτή η επιχείρηση βρέθηκε στην ίδια πτωτική πορεία όπως και η ελληνική οικονομία. Πρόκειται για μια συνεταιριστική επιχείρηση μικρών καταστημάτων που δεν μπορούσε να επιβιώσει και αναγκάστηκε να κλείσει το 2014. Κανένα από τα μέτρα ε, λιτότητος και ιδίως η περικοπή αποδοχών δεν μπόρεσε να το αποτρέψει αυτό. Ε, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε μια σειρά υπηρεσιών στους εργαζόμενους το Φεβρουάριο του 2016 και αυτό πριν από την έγκριση <clears throat> της χρηματοδότησης του Ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Έδωσε ένα προσωπικοποιημένο πακέτο υπηρεσιών στους εργαζομένους, το οποίο έγινε σε συνεργασία με τους ε, κοινωνικούς εταίρους και τους ε, εργαζόμενους και είχε σαν στόχο να αυξήσει την απασχολησιμότητα των εργαζομένων με κατάλληλη κατάρτιση και παροχή ε, δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να έχουν άλλες ε, απασχολήσεις και επομένως ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργαζομένων για να έχουν τις απαραίτητες την απαραίτητη κατάρτιση και τις απαραίτητες δεξιότητες, αυτό είναι το περιεχόμενο του πακέτου, για την, ε, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος να κάνει κάποια σχόλια σχετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ τώρα θα μας πει για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νίριάντα. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό για μας. να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ε, κατάρτιση των εργαζομένων σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν μπορεί πια να λειτουργήσει, να, να συνεχίσει να λειτουργεί η Κομισιόν έχει θεσπίσει το στόχο το 20% του ΑΕΠ να προέρχεται από παραγωγή αγαθών και αυτό μπορεί να είναι η βάση για να μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες ε, στην ε, Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μπορέσουμε τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους για την προστασία του περιβάλλοντος, όσο για τους στόχους παραγωγής να είμαστε φιλόδοξοι και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να τεθεί ο στόχος αυτός και για το 2030, εάν είχαμε το 2020 το στόχο του 20-20-20%, το 2030 θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια παραγωγή η οποία ανακαλύπτει το 30% του ΑΕΠ. Με την επίτευξη αυτών των στόχων θα ξεπεραστούν προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης που δεν έχουν μια επαρκή παροχή ε, αγαθών <clears throat> στους καταναλωτές και αυτό είναι κάτι το οποίο φυσικά θα οδηγήσει σε ανάκαμψη στην απασχόληση στην Ευρώπη και είναι πολύ σημαντικό αυτό να συνοδεύεται από μια διτή εκπαίδευση, διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων και ήδη έχουν ξεκινήσει πολλές πρωτοβουλίες στο θέμα αυτό. Yeah, uh... Ε, Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με όλους όσους λένε ότι το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πολύ περισσότερο Υπάρχουν όμως κάποια κράτη-μέλη και το δικό μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και βρισκόμαστε συχνά σε κατάσταση ε, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές ε, απολύσεις ε, σε χαλιβουργίες, για παράδειγμα, που χρειάζονται πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ βοήθεια. Θα μπορούσε αυτή η βοήθεια να, προ, να προκύψει από το Ταμείο Προσαρμογής, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν κάνει αίτηση. Θα μπορούσαμε έτσι να βοηθήσουμε και την Ελλάδα που έχει οικονομικά προβλήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο θα χρησιμοποιείται από τέτοια κράτη-μέλη. Πολλές φορές ε, ε, εκταμιεύονται τα κονδύλια, αλλά τόσο αργά, καθυστερούν τόσο πολύ ε, που οι άνθρωποι που έχουν απολυθεί έχουν βρει δουλειά αλλού τη στιγμή που θα ε, είναι διαθέσιμα τα κονδύλια από το Τομείο ε, Προσαρμογής Παγκοσμιοποίησης. Ο κύριος Κίρτσος. Και να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την κοινωνική της ευαισθησία. Συμφωνώ απόλυτα με την εισήγησή της. Απλά ήθελα να, να σας πω μερικά πρόσθετα στοιχεία ο, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα περνάει μεγάλη κρίση. Αυτά που εξακολουθούν την προσπάθεια, μεγάλες αλυσίδες, μεγαλύτερες από το Λάρισα σούπερ μάρκετ, βρίσκονται στην ανάγκη να συγχωνευτούν για να επιβιώσουν και έχουν και μεγάλες ε, οφειλές, κυρίως προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγωγούς, ε, αγρότες, ε, κτηνοτρόφους και είναι ένα λεπτό ζήτημα. Επομένως είναι σωστή η παρέμβασή μας ε, προς την κατεύθυνση ε, των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους ε, από το Λάρισα σούπερ μάρκετ και των ανθρώπων που θέλουν ένα νέο ξεκίνημα στην περιοχή. Δυστυχώς η οικονομική προοπτική στην Ελλάδα παραμένει δύσκολη. Το 2015 πήγαμε λίγο πιο πίσω από εκεί που έπρεπε να ήμασταν και το 2016 ε, αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Είναι η αξιολόγηση, ελπίζω να κλείσει θετικά στο άμεσο μέλλον. Ε, πρέπει να επισημάνω όμως δύο προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας ε, του Ταμείου, ε, το οποίο, που δεν έχουν σχέση με εμά, αλλά ε, έτσι επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα μας. Πρώτον υπάρχει η ελληνική γραφειοκρατία που πάντα δημιουργεί κάποια προβλήματα και δεύτερον υπάρχει δυσκολία από την πλευρά των ελληνικών κυβερνήσεων, ιδιαίτερα από το 2015 και πέρα για τη συγχρηματοδότηση, διότι υπάρχει μια διαρκής κρίση ρευστότητας, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους πιστωτές για την αξιολόγηση του προγράμματος. Επομένως, ενώ έχουν εγκριθεί προηγούμενα προγράμματα και με τη δική μου πρόταση, περπατάω στους δρόμους της Αθήνας και βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν πάρει τα λεφτά τους, για παράδειγμα δημοσιογράφοι και τεχνικοί τύπου που έχασαν τη δουλειά τους στα μέσα ενημέρωση στην περιοχή της Αττικής και δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Ε, άρα, ε, συμφωνώ, επαυξάνω, απλά να συνεννοηθούμε ε, και να συνεννοηθούμε και με τις ελληνικές αρχές, ώστε να γίνουν όλα σωστά για να προστατεύσουμε και την αξιοπιστία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Νίριάντα για να συνοψίσει, θα ήθελα να σας υποβάλω έναν προβληματισμό, ερώτηση, στην οποία δεν έχω απάντηση. Η παγκοσμιοποίηση, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη, σε μια πρώτη φάση ήταν επιχειρήσεις ε, οι οποίες εξαφανίζονταν γιατί μεταφερόταν η παραγωγή σε μέρη όπου ε, το ανθρώπινο δυναμικό ήταν φθηνότερο. Μετά υπήρξε ένα πακέτο που αφορούσε τις μεταφορές Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί στερεύλωση ανταγωνισμού εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό, γιατί είναι τόσο διαφορετικές ε, οι νομοθεσίες ε, ε, σε επίπεδο, για παράδειγμα, κοινωνικής κάλυψης, κοινωνικής προστασίας. Είδα σε, στη γαλλική τηλεόραση μια εκπομπή το οδικό, το σιδηροδρομικό δίκτυο της Γαλλίας ε, είχε μεταφέρει ένα τμήμα της ε, παραγωγής της ε, στην Βουλγαρία για να εξελίξει το δίκτυό της και τα φορτηγά κατέληγαν τελικά στην Γερμανία. Στα... Αυτό είναι ένα παράδειγμα για τις για τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε δεσπόζουσα θέση από κάποια ε, σούπερ μάρκετ. Κάποιοι παραγωγοί αναγκάζονταν να μετατοπιστούν για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να ε, αντιμετωπίσουν ε, τους περιορισμούς ε, των σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων σούπερ μάρκετ που πιέζουν τους παραγωγούς να μετατοπιστούν και αυτά τα σούπερ μάρκετ τώρα είναι που αντιμετωπίζουν προβλήματα να τους βοηθήσουμε. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Όταν η μισθωτοί μικρών επιχειρήσεων, μικρών επιχειρήσεων πτωχεύουν ε, ε, υπάρχει ένα θέμα ε, χρήσης του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Τι όμως πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από αυτό το πρόβλημα, κυρία Νηριάντα. Πράγματι αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ορεσμός του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του τι ευελιξία μπορεί να υπάρχει. Γιατί εμείς στην Ιρλανδία έχουμε για παράδειγμα ε, ένα πρόβλημα με την ε, και δεν φταίνει η ίδια ε, φταίνε, φταίει η κατάσταση κάποιων ε, αποθεμάτων. Δεν, φταίνει, δεν φταίει η αλληλεία, φταίει το γεγονός ότι δεν υπάρχει πια το προϊόν που εμπορεύονται. Κάπου υπάρχει ενδεχομένως το ίδιο πρόβλημα και με τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια ευρύτερη συζήτηση, πράγματι, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, πιστεύω ότι πρέπει να την κάνουμε τη συζήτηση κάποια στιγμή σε μεταγερέστερο στάδιο και να συμφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριο. Σεβόν, για το, τη χρονική στιγμή διάθεσης ε, της βοήθειας. Ξέρω ότι σε άλλες χώρες ε, ε, επαφίεται πραγματικά στη διακριτική ευχέρεια από απόψεως συγχρηματοδότησης στα κράτη-μέλη τα ίδια που είναι πολύ συχνά τα ίδια καθυστερούν ε, είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση ε, ανάλογα με το κράτος μέλος. Πρέπει να δούμε πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης από το κάθε κράτος μέλος. Σωστά πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα που να είναι κάποιος πιο περιοριστικό, ώστε να είναι εποφελής η βοήθεια για τους εργαζομένους πράγματι. Κάτι ακόμη ε, το, η ομάδα που πρέπει να, στην οποία πρέπει να στοχεύσουμε πρέπει να καθοριστεί, ακόμη μένει να καθοριστεί. Ε, υπάρχει το θέμα της διευκόλυνσης για την νεολαία και πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Υπάρχουν πάρα πολλά ε, στοιχεία στο Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση που παρουσιάζουν αδυναμίες, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο πρόεδρος. Μάλιστα, να ολοκληρώσουμε αυτό το, αυτή την ανταλλαγή απόψεων για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε σχέση με το σούπερ μάρκετ ε, Λάρισα. Θα ήθελα να πω ότι οι τροπολογίες πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου 12 η ώρα το Μοσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών 23 Μαΐου και η Ολομέλεια θα αποφασίσει στις 25 Μαΐου. Κυρία Νίριαντα, μήπως θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε και το επόμενο θέμα για το οποίο είστε αρμόδια, πώς θα αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μιλάω κατά συρροή ε, τα τελευταία δέκα λεπτά. Πρόκειται για μία ε, έκθεση της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, αφορά την βελτίωση της ποιοτική απασχόλησης και τη δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να δημιουργήσουν καλές και αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης. Ξέρουμε ότι ένα από τα βασικά εμπόδια είναι το πρόβλημα χρηματοδότησης για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα γιατί έχω επιχειρηματικό παρελθόν και ξέρω ότι στην Ιρλανδία αν αρχίσει μια επιχείρηση από το μηδέν και πτωχεύσει ούτε ένα ε, λεπτό του ευρώ δεν μπορούμε να πάρουμε από το κράτος, οπότε δεν πρέπει κανείς να αρχίζει μια επιχείρηση εκτός, εκτός αν είναι απολύτως βέβαιος ότι θα είναι πολύ κερδοφόρα η επιχείρησή του. Ε, είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στήριξη τους, ε, γιατί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη συνοχή και είναι βέβαια η ραχοκοκαλιά κάθε υγιούς οικονομίας όσον αφορά την παραγωγή θέσεων απασχόλησης και Βεβαίω, ε, λόγω τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και στην ένταξη των νέων στην απασχόληση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης ως προς ε, την ε, το, δυναμικό ανάπτυξης της κατάρτισης εντός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ύπαρξης νέων δεξιοτήτων που θα δώσει τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες να αποκτήσουν όλες αυτές τις, τις ε, δεξιότητες από ε, νεαρή ηλικία. Πρέπει να λάβουν υπόψη βέβαια και τις περιφερειακές ανισότητες ε, και η δυνατότητα πρόσβασης και, από τις εθνικές, και στις εθνικές τράπεζες, πιστώσεις εθνικών τραπεζών. Επίσης, μηχανισμός διόρθωσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση όλων των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επικεντρωθούμε κυρίως σε φτωχότερες χώρες ε, και περιφέρειες που αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα και μιλάω για την πρόσβαση ε, των ε, περιφερειών αυτών σε ε, πρόσβαση στη πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των επιχειρήσεων αυτών για την παραγωγή ε, βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και ζητούμε από τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν και το πρόβλημα της απώλειας θέσεων απασχόλησης και να δημιουργήσουν, να συμμετέχουν στη δημιουργία μιας ισότιμης, ενός ισότιμου πεδίου για όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει καμία κρατική εγγύηση. Ε, χρειάζεται λοιπόν πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ξέρω ότι υπήρξαν τροπολογίες στο ESFI που αφορούσε ειδικότερα την κοινωνική οικονομία ώστε να μπορούν οι συνεταιρισμοί να έχουν πρόσβαση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αυτό, ειδικότερα για τις πιο περιφερειακές περιοχές, ε, να μπορούν δηλαδή σε επίπεδο περιφερειακό να δημιουργούν αυτούς τους συνεταιρισμούς και βλέπω τέτοια αποτελέσματα πολύ καλά στην Ιρλανδία, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να υποστηριχθεί. Αυτά είχα να σας πω και αν έχετε ερωτήσεις είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας. Sí, Ευχαριστούμε κύριε Σίδρε. Ο κύριος Ρούμπικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ιδιαίω το θέμα τη δημιουργία θέσεων εργασία θα διαδραματίσει στο μέλλον με μεγαλύτερο ακόμη ρόλο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαίτερα όσον αφορά και την εκπαίδευση. Και το είπα και στο προηγούμενο θέμα για τα σούπερ μάρκετ Λάρισα. Αν δεν καταφέρουμε να ε, ε ενισχύσουμε την παραγωγή στην Ευρώπη και να δημιουργήσουμε και αντίστοιχε θέσει. Ε, εργασίες, δηλαδή 30% έως το 2030, χωρίς τέτοια κίνητρα για την παραγωγή δεν θα τα καταφέρουμε. Και για το σκοπό αυτό χρειαζόμαστε και επιχειρηματίες οι οποίοι θα είναι διατηθειμένοι να αναλάβουν και το ρίσκο, το επιχειρηματικό, να εκπαιδεύσουν και τους υπαλλήλους τους και το ερώτημα που τίθεται είναι τι κίνητρα μπορούν να δοθούν για τον σκοπό αυτό. Αφελώς θα μπορούσα να πω ότι οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει ε, κατέτος να ε, επιτυγχάνουν 1% κέρδος, ε, να υπάρχει ένας τέτοιος κανόνας δηλαδή. Ε, κάτι τέτοιο βεβαίως δεν θα, δε, θα μπορούσε να λειτουργήσει στην, στην πράξη. Ε, θα έπρεπε δηλαδή να, να κάνουμε το αντίθετο. Θα πρέπει να ε, εξασφαλίζεται ε, ότι κάθε επιχείρηση θα έχει μια, ένα επίπεδο κερδοφορίας για να μπορεί να αναλαμβάνει και ευθύνες. Κάτι τέτοιο θα πρέπει και να να επιβραβεύεται. Γι' αυτό και ένας από τους τρόπους θα μπορούσε ε, να είναι να δημιουργηθούν αυτά τα προοδευτικά συστήματα φορολόγησης. Το θέμα που πρέπει να σκεφτούμε όμως είναι ε, που θα το κάνουμε αυτό. Στην, ε, στην, στην Αυστρία, για παράδειγμα, τα πολυτελείας αγαθά δεν φορολογούνται με 20% αλλά με 30%. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική φορολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται και οι πόροι. Για την Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί αυτή η διαδικασία μετεκπαίδευσης. Υπάρχουν ε, προγράμματα ανταλλαγής, προγράμματα ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης ε, μαθητευομένων. Υπάρχουν ε, προγράμματα όπως το Εράσμους για νέους επιχειρηματίες που αυτή τη στιγμή, ε, στο οποίο συμμετέχουν αυτή τη στιγμή 10.000 άνθρωποι στην Ευρώπη. Ενδεχομένως θα μπορούσε αυτό να αναβαθμιστεί και σε διεθνές πρόγραμμα ε, γιατί μόνο αν δημιουργήσουμε επιχειρηματίες οι οποίοι θα είναι διατεθειμένοι να αναλαμβάνουν και επιχειρηματικά ρίσκα, θα καταφέρουμε να οδηγηθούμε και στη δημιουργία θέσεων απασχόλων. Και αυτή είναι η πρόκληση. Ο κύριος Βόν. Ευχαριστώ. Δεν έχει έρθει η σκιώδη των σοσιαλιστών, γι' αυτό μου ζήτησε να πω εγώ ε, εκ μέρους της κάποια, ε, λόγια. Ε, καταρχάς να συγχαρώ τον, τον εισηγητή, την εισηγήτρια μάλλον για την έκθεσή της, ιδίως για το γεγονός ότι περιλαμβάνονται προτάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε την ανάπτυξη αυτών των, ε, ε, την, ε, επιχειρήσεων. Θέλουμε οι μικρές να γίνονται μεσαίες και οι μεσαίες να γίνονται μεγάλες. Έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Επίσης, σημαντική είναι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης δεν ε, δεν είναι καν γνωστή σε πολλές ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, για παράδειγμα, έχουν διευκολυνθεί κάποιες διαδικασίες. Υπάρχει ένα ποσοστό τον, το οποίο θεωρούμε εμείς ότι θα πρέπει να δαπανάτε για, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι υπάρχει και μια τέτοια πρόθεση για τα επόμενα χρόνια. Με όλα αυτά ε, πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η, τα προγράμματα ε, εκπαίδευσης και έτσι θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από αυτά τα ταμεία. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα και νομίζω ότι θα πρέπει να δίνονται ευκαιρίες ε, και μέσω του ε, χρηματοδοτικού μέσου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως. Και πολλές ε, επιχειρήσεις, παρότι πολλές φορές γνωρίζουν ή και δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, πολύ λίγες γνωρίζουν πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να χρηματοδοτηθούν από τα ε, μέσα αυτά. Και πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για ε, να διαφημίσουμε αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποβάλουν αιτήσει για χρηματοδότηση. Αυτές είναι ευκαιρίες που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά και πραγματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Νοβάκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Νιράντε, γιατί είναι πολύ εξισορροπημένο το έγγραφο που μας παρουσίασε. Εγώ ως εισηγητής, ε, ως ε, συντάκτης νομοδότης Επιστροπής ε, ε, περιφερειακής ανάπτυξης, θα ήθελα να ε, μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες και γι' αυτό ε, έχω συμπεριλάβει, θα ήθελα να συμπεριληφθούν πολλά σημεία της γνωμοδότησης όσον αφορά τις εγγυήσεις, τις μικροπιστώσεις, γιατί για την ώρα έχουμε περισσότερα χρήματα από, καλές, από ότι καλές ιδέες για το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή έχουμε ε, διαθέσιμους πόρους, ο κόσμος δεν ξέρει πού να πάει και τι να ζητήσει, οπότε είτε πηγαίνουν στις τράπεζες για να πάρουν ένα τραπεζικό δάνειο και να πληρώνουν υψηλό ε, τόκο αποπληρωμής ή... Ε, προσπαθούν να ε, συμμετέχουν σε διάφορα project με ε, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα εγχειρίδιο κανόνων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν περισσότερο όσον αφορά την χρηματοδότηση της Ένωσης. Πρέπει να επικεντρωθούμε στις χώρες που απορροφούν ε, σε πολύ χαμηλό βαθμό την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί Αυτές οι, αυτές οι περιφέρειες ε, ε, δεν έχουν το δυναμικό να τα αξιοποιήσουν. Πρέπει να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτές. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προοδεύσουν όσον αφορά την απλοποίηση της ε, χρηματοδότησης της Ένωσης από το μηχανισμό υποβολής αιτήσεων μέχρι τον έλεγχο. Και όταν μιλάω για έλεγχο, λέω ότι ο έλεγχος πρέπει να γίνεται επί τη βάση αξιολόγησης κινδύνου. Οι χώρες που έχουν πολύ καλό ιστορικό πρέπει να ε, είναι αντικείμενο λιγότερης, ε, λιγότερο ελέγχων και να ε, έχουν να αντιμετωπίσουν λιγότερη γραφειοκρατία, ενώ οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρέπει να ελέγχονται περισσότερο για να μην υπάρξει κίνδυνος κατάχρησης όσον αφορά το κόσμο και τον ορίζοντα 2020. Είπα και στο παρελθόν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν 55 εκατομμύρια ε, που τους έχουν διατεθεί για 5 χρόνια. Είναι ελάχιστο, είναι, είναι πάρα πολύ ε, χαμηλό αυτό το ποσόστο για 28 ε, χώρες. Οπότε χρειάζεται μία συζήτηση εκτενής στο Κοινοβούλιο το 2006 για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Εμείς ζητούμε μακροχρόνιες πολιτικές για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ε, στόχους και αυτό το ζητούμε από τα κράτη-μέλη, αλλά εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά το 2020. Οπότε όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρων, αναχώρες, ε, αναχώρα, πρέπει να τις συνδέουμε με το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ε, δεν πρέπει να γίνεται να υπάρχει κανονιστικός υπερθεματισμός στα κράτη-μέλη, γιατί αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Ε, όταν πηγαίνουμε σε κάποιο δικαιούχο σε μια χώρα ε, και τον ρωτάμε, δεν ξέρει ότι υπάρχει ένα μέσο ή ένα τρόπο υποστήριξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση για μια μικρομεσαία επιχείρηση. Κάτι ακόμη ε, όταν υπάρχει μια μεγάλη κρίση δεν πρέπει να ε, μειώνονται οι δυνατότητες παροχής κονδυλίων στο πλαίσιο του στόχου 3. Δηλαδή όταν υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όπως το προσφυγικό για παράδειγμα. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία για να φύγουν τα χρήματα από τον ορίζοντα 2020 ή από το κόσμο για να πάνε στο, ε, στην προσφυγική κρίση. Δεν θα μ' άρεσε η Ευρωπαϊκή μας Ένωση ε, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή, όταν θα έχει περάσει αυτή η κρίση, εντάξει, όχι τη Δευτέρα που μας έρχεται, αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτή η κρίση, δεν, θέλουμε να, δεν θέλω να μην υπάρχει κανένα απολύτως, καμία χρηματοδότηση ε, για άλλα, άλλους στόχους και άλλες προτεραιότητες που έχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεβανόη, τελευταίος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κινείται προ την σωστή κατεύθυνση η έκθεση. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία ιδιαίτερα. Καταρχήν για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε απομονωμένες περιοχές. Είναι μια πραγματικότητα και αυτή. Το να είναι κάνει σε μια περιοχή της υπαίθρου, ιδίως ε, απομονωμένη, θίγει τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στι υποδομές, οι οποίες υποδομές δεν υπάρχουν σε απομονωμένες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει πολιτική θέληση για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στον αγροτικό χώρο, γιατί εκεί πραγματικά υπάρχουν μεγάλες ανισομέρειες στις επικρατείες μας. Μια δεύτερη πτυχή, το θέμα των ε, κοινωνικών ενώσεων και των συνεταιριστικών ενώσεων που αναφέρθηκαν στην έκθεση αυτή. Πρέπει να αντιμετωπίζονται οι συνεταιριστικοί οργανισμοί με διαφορετικό τρόπο, με τον ίδιο τρόπο από ότι οι υπόλοιπε επιχειρήσει, κάτι το οποίο δεν γίνεται ακόμα σήμερα. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπαμε σήμερα για την παγκοσμιοποίηση. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να προβλέψουν και να προκαταλάβουν αυτά τα οποία θα γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο και θα είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση να τις βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτή είναι μια ε, πρόταση που καταθέτω στην ε, έκθεσή μου για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Πρέπει να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να καταλάβουν τι έρχεται και να προετοιμαστούν με τις απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Ευχαριστούμε την κυρία Νάρια Νίριαντά που θα κλείσει τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ όλους <clears throat> για, την, ε, για τις παρεμβάσεις σας είσαστε καλόδεκτοι να μου πείτε αν θέλετε κάποια τροποποίηση στην έκθεση αυτή. Έχουμε ακόμα κάποια πρόσθετα στοιχεία που μπορούν να συμπεριληφθούν στην έκθεση αυτή. Και σίγουρα μπορείτε να συνδέσετε και αυτή την έκθεση με την προηγούμενη έκθεση που παρουσίασε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Γιατί συνδέονται. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε για το πρόβλημα τη πληροφόρηση. <clears throat> αυτό όμω είναι ένα γενικό πρόβλημα στην Επιτροπή Προπολογισμών δεν είναι μια τόσο γητευτική και συναρπαστική επιτροπή. Νομίζω ότι ο κόσμος όταν τους λέτε για χρηματοδοτικά εργαλεία πάει το μυαλό του στα μουσικά όργανα, τα instruments στα αγγλικά, financial και musical. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι σας είσαστε στην ίδια κατάσταση με μένα όταν πηγαίνω στην εκλογική μου περιφέρεια στο Κέννη, στην Ιρλανδία, τους ενδιαφέρει πώς θα βρούνε μέσα χρηματοδότησης. Δεν θέλουν να κάθονται και να τα ψάχνουν ήδη. <clears throat> Επομένως το θέμα είναι να παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση και να βοηθούμε τις εταιρείε οι οποίες έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους στο παρελθόν και να μην τις βάζουμε κάτω από ένα γραφειοκρατικό ζυγό, αλλά παρόλα αυτά και τις νεοφύης επιχειρήσεις να τις βοηθήσουμε. Όλα αυτά τα λέω στην εκθεσή μου για τις συνεταιριστικές εταιρείε. Πάντα λέω, ήμουνα σε μία από τις ε, πόλεις στην Ελλανδία που κλείαν όλα τα μαγαζιά, όλο και περισσότερο. Και είχα την εξή ιδέα, υπήρξε ένα μαγαζί που είχε τρεις ε, ιδιοκτήτες που κάναν τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις στον ίδιο χώρο, ένα βιβλιοπωλείο, ένα ραφτάδικο και ένα ακόμα που πουλούσε, ένα μαγαζί που πουλούσε μουσικά όργανα και μπορούσαν έτσι να μειώνουν το κόστος της ε, <clears throat> ενοικίασης και της φορολογίας με το να έχουν κοινό χώρο εμπορίας και έτσι βοηθούσαν και τους ανθρώπους που ερχόντουσαν να πάρουν κάτι παραπάνω από τον καθένα. Είναι αυτό λοιπόν μια καινοτόμα ιδέα η οποία μπορεί να ενθαρρυνθεί και για μένα που έρχομαι από μια αγροτική περιοχή της Ιρλανδίας. Ο στόχος μου είναι να δώσουμε και πάλι αναζωγόνηση της ε, αγροτικής οικονομίας και να πάρει την απαραίτητη αυτονομία ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και να δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Εγώ προσβλέπω λοιπόν στην συμπλήρωση αυτής της έκθεσης <clears throat> και αν έχετε κάποια ερωτήματα παρακαλώ να απευθυνθείτε σε μένα. Κάτι ακόμα για αυτούς που, που δεν ξέρουν να προφέρουν το όνομά μου. Λέγεται με Λία. Αυτό αρκεί. Ευχαριστώ Λία λέει ο πρόεδρος παρά την αριστεία της έκθεσης αυτής, ενδεχομένως θα υπάρξουν τροπολογίες. Εάν προκύψουν τροπολογίες, πρέπει να κατατεθούν μέχρι 28 Απριλίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει στις 23-24 Μαΐου. Και η Επιτροπή Απασχόλησης θα αποφασίσει στις 15 Ιουνίου, γιατί αυτή είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Παραμένουμε στις μικρομεσαίες τώρα και την πρόσβασή τους στην αγορά κεφαλαίων. Έχουμε τώρα τον κύριο Κούσμιουκ, ο οποίος είναι εισηγητής για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Υπόθηκαν πολλά για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην προηγούμενο, στο προηγούμενο θέμα και για το κάθε κράτος μέλος ε, ξεχωριστά αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Εγώ θα επικεντρωθώ στο ζήτημα της ε, χρηματοδότησης. Η γνωμοδότηση που έχω συντάξει απευθύνεται στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Οι προτάσεις μας, λοιπόν, είναι λίγες. Να σας επισημάνω το γεγονό ότι όσον αφορά την εξωτερική χρηματοδότηση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χρηματοδοτούνται κατά 80% από τράπεζες και μόνο κατά 20% από κεφάλαια αγορές. Και η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ε, δυσκόλεψε πάρα πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το να αποκτήσουν πρόσβαση σε δάνεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως βεβαίως και το ΕΤΣΕ. Δεν θα σας ε, παρουσιάσω ολόκληρη τη γνωμοδότηση, παρά μόνο κάποια σημαντικά στοιχεία που αποτελούν τη βάση της. Πρώτον, ήθελα να τονίσω ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διευκολύνει περισσότερο την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγορές και σε χρηματοδότηση. Να τονίσω επίσης ότι τα προγράμματα υποστήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον έως το τέλος του τρέχοντος πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Επίσης, τονίζω τη σημασία των προσπαθειών που πρέπει να κάνουμε για τη διατήρηση του προγράμματος COSME. Επίσης, γράφω ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δόθηκαν 75 ε, δισεκατομμύρια ή χορηγήθηκαν 75 δισεκατομμύρια από το EFSI σε αυτόν τον κλάδο της οικονομίας και θα παρακολουθούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις ε, αυτής της ε, κίνησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ε, αυτό, είναι πολύ αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ιδίως για τις φτωχικότερες περιοχές, είναι η γεωγραφική κατανομή της χρηματοδότησης. Επίσης υπάρχει μια... αναφέρω ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί πλήρως η ρήτρα ευελιξίας. Επίσης, λέω ότι χαιρόμαστε πολύ που τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία ε, ε, έχουν ανοίξει περισσότερο προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τονίζω ότι εμείς υποστηρίζουμε τη μετακίνηση από τις επιχορηγήσεις προς τις εγγυήσεις γιατί στρεβλώνουν λιγότερο τον ανταγωνισμό. Επίσης τονίζω το, τη σημασία των διαρθρωτικών ε, ταμείων της διαρθρωτικής χρηματοδότησης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Και τέλος αναφέρω τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Θεωρούμε, θεωρώ ότι θα πρέπει να εμ, και να καταστούν πιο ευέλικτοι οι σχετικοί κανονισμοί και οι σχετικοί κανόνες. Εμείς, αν έχετε ε, κάποιες ιδέες για τροπολογίες, μπορείτε να τις υποβάλλετε μέχρι τις 20 Απριλίου. Ευχαριστώ, Λεοπρόεδρος. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα, λέει ο κύριος Ρούμπικ. Γνωρίζουμε ότι ξεκινούμε πάντα με τη διαπίστωση ότι κάποιος ο οποίος είναι αυτοαπασχολούμενος κάνει ένα μεγάλο ε, άλμα, το, είναι το πρώτο άλμα που κάνει κανείς προς το επιχειρήν, συνοδεύεται από μεγάλο κίνδυνο. Και φυσικά πολλοί αυτοαπασχολούμενοι κάνοντας αυτή τη μετάβαση αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή Προϋπολογισμών να προετοιμαστεί για το, την επιχειρηματική δράση για τις γυναίκες επιχειρηματικούς αγγέλους διότι οι γυναίκες χρειάζονται πολύ περισσότερη ευελιξία στον επιχειρηματικό χώρο και προγράμματα όπως αυτό για τις γυναίκες αγγέλους το βελτιώνουν και το ευνοούν. Έχουμε εγκρίνει ένα πρόγραμμα λοιπόν για το επιχειρήν το οποίο είναι και πρόσφορο στο να αντιμετωπίσει την ε, απασχόληση των ε, μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι έχουν έρθει ένα εκατομμύριο ήδη στην Ευρώπη. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ε, μετανάστες να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι και επίσης μπορούν να απασχολήσουν και ε, συντοπίτες τους οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες γλωσσικές γνώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινότητός τους. Είναι απαραίτητο επίσης να τονίσω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνέχεια ζητά να μάθουν περί τίνος πρόκειται και τι δυνατότητες έχουν, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τις απαραίτητες χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Σας καλώ λοιπόν να σκεφτείτε και εσείς πώς μπορούμε στο ορίζον 2020 να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενδεχομένως και με μεταφορές πιστώσεων σε ορισμένες θέσεις, γιατί εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια διαδικασία που θα οδηγήσει σε περισσότερη ανάπτυξη του τομέα αυτού. Έχουμε λοιπόν τις απαραίτητες γνώσεις, έχουμε την οργάνωση που χρειάζεται, αλλά θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνει όλη αυτή η δραστηριότητα σε ευρύτερους και ευρύτερους χώρους. Είναι οι μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν τις θέσεις εργασίας, όπως γνωρίζουμε όλοι, και εκεί θα βρεθούν οι νέες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή την ανάπτυξη του τομέα αυτού που μπορεί να είναι σημαντική. Ο κύριος Βόν. Ε, ευχαριστώ πολύ. Η Κλέρη και η μας, δεν είναι εδώ. Ούτε το γονατό θα ήθελε όμως ε, να ευχαριστήσει τον εισηγητή. Δεν είναι όμως ε, μία έκθεση με την οποία θα συμφωνούσαμε. Θα συμφωνούσαμε με τη σημασία του κόσμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε καλύτερους τρόπους διαφήμισης αυτού του μέσου, ώστε να γνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι υπάρχει και πώς πρέπει να υποβάλουν έτοιμοι. Επίσης, συμφωνούμε με το γεγονός ότι 75 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, όμως θα θέλαμε στο μέλλον να το παρακολουθήσουμε αυτό, να δούμε ότι όντως αξιοποιούνται τα κονδύλια αυτά από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και αν ε, ήταν αποτελεσματικά από απόψε ως δημιουργίας επιχειρήσεων αλλά και θέσεων απασχόλησης. Όλοι θα συμφωνούσαμε με τη δήλωση ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ένωσης πρέπει να είναι απλούστερη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν πηγαίνω σε επισκέψεις ε, ε, με ε, την Επιτροπή μας και συναντούμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας λένε συνεχώς ότι οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλούστεροι για εκείνες. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία λοιπόν μεταξύ της εξασφάλισης του γεγονότος ότι είναι άμεσα προσβάσιμα τα ε, κονδύλια για μικρότερα projects ή για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά να εξασφαλίζουμε επίσης ότι τα χρήματα ε, αξιοποιούνται σωστά. Είναι δύσκολη αυτή η ισορροπία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν μπορέσουμε να την καταφέρουμε, νομίζω θα είναι καλό. Επίσης, ε, η ομάδα υψηλού επίπεδου για την απλοποίηση, για την απλοποίηση ξέρω ότι έχουν κάνει κάποιες πρώτε συζητήσει για κάποιες πρώτε προτάσεις. Ε, θα είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να υπάρξουν ιδέες ε, για την απλοποίηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το διερευνήσουμε. Για το σημείο 5 ε, ο εισηγητής αναφέρεται στη μετατόπιση ε, από τις επιδοτήσεις, τις εγγυήσεις ή τα δάνεια. Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός είναι όλο και μικρότερος, είναι πώς θα χρειαστεί αυτό, θα χρειαστεί να ε, εξαρτώμαστε περισσότερο από δάνεια και εγγύησεις, αλλά ίσως θα έπρεπε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε κάποιου είδους επιδοτήσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή σε μικρότερα projects, απλώς ε, αρκεί να μην κάνουν αίτηση και ε, σε άλλου είδους ε, ταμεία. Πρέπει λοιπόν να το αποδεχθούμε αυτό, ότι θα υπάρξει αυτή η μετατόπιση, όμως δεν πρέπει να εξαφανιστούν εντελώς οι δυνατότητες υποβολής αιτήσεων για επιδοτήσεις, τουλάχιστον για τα μικρότερα projects. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κύριε Σιγητά, έχετε παρατηρήσεις. E, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις σας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τις δικές μου σκέψεις, όπως εκφράζω στην γνωμοδότησή μου και συμμερίζομαι την άποψή σας ότι είναι απαραίτητη η αύξηση της χρηματοδότησης για τον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό θέλουμε. Ε, πρόκειται για ένα από τα βασικά θέματα της γνωμοδότησής μου. Και ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα είναι ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν οι επιδοτήσεις με εγγυήσεις προκειμένου να υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης του κλάδου από τον προϋπολογισμό και επίσης τονίζουμε στην γνωμοδότηση το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για τον συγκεκριμένο ε, κλάδο. Αυτά τα 75 δισεκατομμύρια του ε, EFSI θα μπορούσαν ακόμη και να αυξηθούν και κάτι τέτοιο μπορεί να ε, βελτιώσει την ανάπτυξη της, ε, του, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να υποβάλλετε τροπολογίες, αν και δεν υπάρχει πολύ χρόνος. Ναι, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι στις 2 Μαΐου στις 18 το απόγευμα. Συγγνώμη, στις 28 Απριλίου λέει ο πρόεδρος. 28 Απριλίου το μεσημέρι. Η ψηφοφορία 23-24 Μαρτίου Μαΐου, συγγνώμη, και η Επιτροπή ΕΚΟΝ, η οποία είναι η αρμόδια επί της ύλης, 13-14 Ιουνίου θα ψηφίσει και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη χρηματοδότησή τους. Ξέρετε ότι το απόγευμα θα έχουμε μια συζήτηση, μια ακρόαση, ε, όπου θα, θέλετε, θα θέλατε ίσως να ε, συμμετάσχετε και η οποία έχει προταθεί από την συνάδελφό μας την Λία. Και τώρα. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη γνωμοδότηση, για την έκθεση πρωτοβουλίας για την ε, πολιτική, εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, που είναι ο υποφαινόμενος. Η έκθεσή μου είναι μια έκθεση κριτικού χαρακτήρα, που εκφράζει ανησυχίες και εκφράζει τη λύπη της, γιατί τίθεται το θέμα της ε, αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <clears throat> Θέλουμε να έχουμε μια <clears throat> κοινή πολιτική εξωτερικών θεμάτων και ασφάλειας, αλλά αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι έχουμε μονάχα περίπου 320 εκατομμύρια, δηλαδή 0,2% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αμυντικά και ασφαλιακά θέματα. Και αυτός ο προϋπολογισμός υποχρησιμοποιείται. Μονάχα 96 εκατομμύρια χρηματοδο... χρηματοδοτήθηκαν από το μάλλον 196 εκατομμύρια. Αυτό δείχνει μια έλλειψη φιλοδοξίας, μια ζωφερή πραγματικότητα μέσα στην οποία βρίσκονται οι Ευρωπαίοι όταν οι διεθνείς συγκρούσεις απειλούν την ασφάλειά μας, την ασφάλεια της Ευρώπης πέραν των στρατιωτικών ε, επιχειρήσεων κατά των διακινητών στην ε, ε, Μεσόγειο και την ενέργεια για το ΚΑΠ Σαχέλ, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Σαχέλ. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη μεταναστευτική κρίση είναι πάρα πολύ περιορισμένη και δεν διατρέχεται από μια πραγματική στρατηγική και σε μια εποχή ε, <clears throat> έλλειψης πόρων στον προϋπολογισμό και ενώ έχουν μειωθεί οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη εναντί άλλων περιοχών του κόσμου, τα κρατη ακόμα δεν καταλαβαίνουν την ανάγκη να επιτύχουν οικονομίες κλίμακος με διαφθορτική και μόνιμη συνεργασία στα αμυντικά θέματα, όπως προβλέπει και η συνθήκη μας, δηλαδή να μπορούν να τίθενται από κοινού τα διάφορα ε, ε, οι διάφοροι στρατιωτικοί πόροι, όπως λέγεται και στο άρθρο να, να τονιστεί ο ρόλος των σχηματισμών μάχης των battle groups και καταδικάζω το γεγονός ότι λόγω της πολυπλοκότητας του σχήματος και είναι παράδοξος ο τρόπος της χρηματοδότησής τους, δεν υπάρχει πραγματική και σωστή χρήση των ε, σχηματισμών μάχης, κάτι το οποίο μπορεί να υπονομεύσει και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι δυνατότητε που παρέχονται από τι συνεργασίε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση από τα κράτη-μέλη και επίση ανησυχώ και για το πάγωμα του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Αμυντικού Φορέα μετά από το 2010 θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κινητοποιηθούν οι δυνατότητες έρευνας στον τομέα της ε, άμυνας ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να προετοιμάσουμε καλύτερα το μέλλον. Είναι απαραίτητο να υπάρξει και ένα πιλωτικό σχέδιο και υποστηρίζω το σχέδιο του Κοινοβουλίου. Από το 2017 θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι οι οποίοι να ξεπερνούν τους πόρους που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει για άλλα πιλωτικά σχέδια και προπαρασκευαστικές δράσεις. Τούτου λεχθέντος, δίνω το λόγο στον κύριο Γκονσάλες Πέρες τώρα. Να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την άψογη εργασία του σε αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι ένα πολύ καλό έγγραφο εργασίας, είναι σύντομο, εξισορροπημένο και καλύπτει τα κύρια σημεία του προβλήματος αυτού. Με το κείμενο αυτό λοιπόν, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μπορεί να εκφράσει την ικανοποίησή της και η Επιτροπή μας, η Επιτροπή Προϋπολογισμών επίσης. Για μένα είναι ενδιαφέρον το ότι λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος που διατρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κρίση των προσφύγων και την ε, απειλή των τζιχαδιστών τρομοκρατών και η ανάγκη να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει την κατάλληλη χρηματοδότηση για την πολιτική ασφάλεια και εξωτερικό θεμάτων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια μόνιμη διαφορεμένη συνεργασία, γιατί αυτό είναι από τα κύρια εργαλεία τα οποία έδωσε τον εαυτό τη μέσα τη συνθήκη τη Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά που μέχρι στιγμή δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώ και υλοποιηθεί. Θα θέλαμε στον υπόλοιπο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου να θίξω και το θέμα της ναυτικής ε, επιχείρησης στη Μεσόγειο, ιδίως με την πρόσφατη πρόοδο που έχει επιτευχθεί με τις ε, λυρικές αρχές. Είναι μια ενέργεια που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη και έχει διασώσει ήδη 3.000 μετανάστες. Θα έπρεπε επίσης να αναφερθεί και το θέμα των καταπιστευμάτων, των trust funds, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τύχη των καταλήλων υποσχέσεων από τους χρηματοδότες και δεν υπόκεινται αυτή τη στιγμή σε επαρκή έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τη χρήση αυτών των κονδυλίων. Στις 27 Απριλίου θα γίνει μια συγκεκριμένη συνεδρίαση μεταξύ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εκεί θα συζητηθούν τα θέματα αυτά. Οπότε επιφυλάσσουμε τις τελικέ μου θέσεις μέχρι να γίνει αυτή η συνεδρίαση, λέει ο κ. Σας Σα ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε κύριος Ντεσόφσκι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να σας, ευχαριστη... να σας ε, ευχαριστήσω και εγώ γιατί η γνωμοδότησή σας αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Εμείς προσκεκλήθημεν ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ένατη Σύνοδο Κοινοβουλευτικών της Ασίας και της Ευρώπης, στη διακοινοβουλευτική αυτή σύνοδο και μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Τσαρνέσκι εμείς εκπροσωπήσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά υπήρχαν και εκπρόσωποι διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών και κοινοβουλίων. Στην Μογγολία όμως δεν υπήρξε καμία, δεν υπάρχει καμία εκπροσώψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στα νησιά Φίτζη, έχουμε μια πρεσβεία. Προσπαθούμε να κάνουμε γνωστά τα συμφέροντά μας εκεί. Στην Μογγολία <clears throat> όμως δεν έχουμε την κατάλληλη εκπροσώπηση. Δεν υπάρχει παρουσία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αναρωτιέμαι λοιπόν κατά πόσο η κοινή προμήθεια στρατιωτικού υλικού δεν θα πρέπει να γίνεται να γίνεται από κοινού. Γιατί παραγωγής χάρη η τσεχική δημοκρατία θα πρέπει να αγοράζει στρατιωτικό υλικό με καλύτερες συνθήκες από ότι η Πορτογαλία ή άλλες χώρες. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε κοινό στρατό, Ίσως θα μπορούσαν να πιστούν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει μια ορθολογικοποίηση των δαπανών των στρατών, που είναι βέβαια πολύ διαφορετικές από τη μια χώρα στην άλλη. Μια τέτοια ορθολογικοποίηση θα πρέπει να συνεχιστεί και αυτό ήθελα να τονίσω. Ευχαριστώ, Ρίκιο Πρόεδρος. Ε, κυρία Μούντι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον ε, συντάκτη της νομοδότησης. Η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας έχει μια σειρά από δυνατότητες ε, χρηματοδότησης αναπτυξιακών πολιτικών, πολιτικών άμυνας, πολιτικών ασφάλειας που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων, ε, που θα μπορούσαν να συμπληρώνουν και το έργο του ΝΑΤΟ και όπως είπα έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα η πολιτική αυτή. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές όσον αφορά το τι μπορούμε να επιτύχουμε τελικά μέσω αυτής της πολιτικής. Πολλές χώρες ε, δεν θεωρούν ότι αυτή η κοινή χρήση των πόρων ε, θα ήταν θετική. Και αυτό αφορά και τη δική μου χώρα βέβαια. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί όσον αφορά το σχεδιασμό και την, ε, και την γρήγορη ανάπτυξη των πόρων που έχουμε στην ε, διάθεσή μας με τον βέλτιστο τρόπο. Ε, θεωρούμε ότι χρειάζονται έξυπνες αποστελές που θα αξιοποιούν τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση κρίσεων και θα ενισχύουν την συνεργασία. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ αυτού οι οποίοι εκφράστηκαν. Ο κύριο Γκονσάλε Πόν μα τόνισε τη σημασία τη ναυτική επιχείρηση στη Μεσόγειο. Βέβαια, μέσω και της ε, Frontex υπάρχει σημαντική συνεισφορά ε, του Ιταλικού ναυτικού όταν ε, σαλπάρουν τα πλεούμενα από τις ακτές της Λιβύης, η Frontex καλύπτει τις ε, ε δαπάνες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις, ε, το στόλο αυτό των διακινητών. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια λακωνική αναφορά σε όλα αυτά. Ουσιαστικά είναι απλώς ε, μια χειρονομία συμβολική. Έχουμε ένα προϋπολογισμό που μόνο κατά τα δύο τρίτα αντιμετωπίζει, μόνο κατά τα δύο τρίτα εκταμιεύεται. Έχουμε δυνατότητες οι οποίες δεν έχουν κινητοποιηθεί και των οποίων η κινητοποίηση θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Το σύστημα κατανομής στο πρόγραμμα Ατενά είναι άδικο γιατί βαραίνει ιδίως τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν την Προεδρία του Συμβουλίου κάθε, κάθε φορά και επομένως πρωτού ξεκινήσουν μπορεί να έχουν σημαντικούς διστάγμους και έτσι το σύστημα Ατένα δεν οδηγεί σε τίποτα. Δίνουμε λοιπόν την εικόνα και την εντύπωση ότι έχουμε μια ικανότητα, αλλά αναρωτιούνται όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες τι κάνει η Ευρώπη και βλέπουν ότι η Ευρώπη βρίσκεται στην αδράνεια και στην αδυναμία δράσης. Αυτό ουσιαστικά δίνει έφορο έδαφος σε όλους τους ξενοφόβους και τους λαϊκίστες. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό μας και να πάρουμε και απαντήσεις από το Συμβούλιο. Επίσης για τον επιμερισμό των προμηθειών στρατιωτικού υλικού και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και επίσης για το θέμα και των ε, διπλωματικών εκπροσωπήσεων. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα μπορούσαμε εμείς ως Επιτροπή προϋπολογισμών να σταθούμε και στις προτάσεις για την αγορά ακινήτων στις, στην, από την υπηρεσία εξωτερικού, εξωτερικής δράσης. Ε, μπορούμε να μοιραστούμε κτίρια μεταξύ κομισιών και κοινοβουλίων σε πόλεις όπως είναι το Πεκίνο ή το Τόκιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε οικονομίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ξεπερνάω βέβαια ίσως το έδαφος ξεπερνώ την οριακή γραμμή για την εθνική κυριαρχία αλλά έχουμε δει και ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επενέβησαν στη Λιβύη και τη Συρία, οδήγησαν στην ε, καταστροφή του κράτους εκεί, κάτι το οποίο οδήγησε σε τεράστια μετανάστευση από τις περιοχές αυτές προς την ε, προς την ε, Ιταλία και την Λαπεδούσα. Σε πολλές, πολλές περιπτώσεις λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται μια επέμβαση, μετά οι Αμερικανοί βγάζουν την ουρά τους και ακολουθούν οι μεταναστεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα μέχρι τις 2 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Είναι η προθεσμία στις τροπολογίες, 23-24 Μαΐου θα ψηφίσουμε και η Επιτροπή η οποία είναι αρμόδια Επί της ουσίας η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει στις 14 Ιουνίου. Ομιλών διαψήφους θα περάσω στην διαδικασία ψηφοφοριών. Παρακαλώ, θέσατε τις κάρτες σας στην αρμόδια σχισμή να ελέγξουμε αν λειτουργεί το σύστημα. Άρχεται η δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψήφιστε όπως θέλετε. Κάποιοι λείπουν ακόμα, κάποιοι δεν. 26 κάρτες, 23 μονάχα έχουν ψηφίσει, 28 τώρα. Bon, τη ε, ψηφοφορία.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 ψήφους έχετε στη διάθεσή σας. Είστε τέσσερις. Κάποιος από εσάς θα πρέπει να μην ψηφίσει. Εντάξει, αποφασίσατε, ωραία. Λοιπόν, πρώτο έγγραφο που θα ψηφίσουμε δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικός έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 15 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι κατά. 14 έχει αποσυρθεί, 15 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 ψήφοι κατά, 13 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 15-13-1. 20 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρας απορρίπτεται. 15 ψήφοι υπέρ και, ε, κατά συγγνώμη και μία αποχή. Πάμε στην τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται 15 ψηφί κατά 13 υπέρ. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Έναρξη. Πέρασα. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 10 κατά και 2 αποχές. 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της τροπολογίας 25. Έναρξη. Πέρασε. Πέρας. 14-14. Άρα απορρίπτεται. 5. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος και πάλι. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρασε. Εγκρίνεται. 16-13. Τροπολογία 26. Υπέρ. Α, καταπίπτει, συγγνώμη, συγγνώμη. Τροπολογία 27. Υπέρ. Α, και, αυτός, και αυτή καταπίπτει. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται 13 ψήφοι κατά 12 υπέρ, 4 αποχές. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Α, καταπίπτει. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος της 29 υπέρ, ε, συγγνώμη, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται 17 κατά 11 υπέρ. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου που τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, έναρξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται 25 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πάμε τώρα στο Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αφρική. Κυρία Γκάρτια Ζαμπάλ. Και της κυρίας Γκάρτια Ζαμπάλ. Συμβεβαστική Α. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Έναρξη ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία υπαριθμών 4. 17 με 11 και μία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Σε. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική δε υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο του κειμένου με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν υπάρχουν ε, αποχές. Ε, ευχαριστώ και συγχαίρω και την εισηγήτρια κυρία Γκουαρδιά Σαλ. Το σχέδιο για τον έλεγχο του Μητρώου των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ναι, ναι, συγγνώμη. Έχουμε προηγουμένως η έκθεση το σημείο 13 θα έρθει στο τέλος μετά από αυτά που ζήτησε η συγκίτρια είναι το λόγο στο Ζωζέ Μανουέλ Δεν έχετε καθόλου μεταφορές. Ο Ζεράν Ντεπρέ για τις μεταφορές τους άλλους τομείς, μεταφορές πιστώσεων στους άλλους τομείς. Ναι κύριε Πρόεδρε κανένα πρόβλημα. Η πρώτη μεταφορά αφορά το ελεκτικό συνέδριο σε δύο σκέλη. Πρώτον, μία αλλαγή σε μία, μία θέση Α σε θέση AD5 μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του ελεκτικού συνεδρίου και επίσης μια μεταφορά πιστώσεων 85.000 ε, ευρώ για να καλυφθεί η ανάγκη της ε, των αμοιβών επί τη βάση της αλλαγής των ελάχιστων μισθών στο Λουξεμβούργο. Δεύτερον, κοινή αίτηση της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 110.000 ευρώ που δίνονται από την Επιτροπή των Περιφερειών 290 από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για να καλυφθούν οι ανάγκες σε επίπεδο ενέργειας και απόδοσης περιβάλλοντος, κάτι το οποίο θα το εγκρίνετε όλοι φαντάζομαι, και για να αντιμετωπιστεί η γύρανση, η τεχνική γύρανση των εγκαταστάσεων των δύο Ελπίζω δεν έχετε καμία αντίληση, εγώ προσωπικά δεν έχω. Αν δεν υπάρχουν αντίλησει, δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε, εγκρίνονται αυτές οι μεταφορές πιστώσεων. Δεν θέλει κανείς να ψηφίσει. Λοιπόν, υπάρχει ένα κείμενο που ήρθε καθυστερημένα σε σχέση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Δεν βλέπω όμως να είναι πρόβλημα. Το ένα αφορά την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το άλλο την Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά και η κοινή πολιτική και για τα δύο όργανα, γιατί έχουν κάποιες κοινέ εγκαταστάσεις. Κανονικά πρέπει να επιφυλαχθούμε λόγω της καθυστέρησης, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη να ψηφίσουμε, μπορούμε να εγκρίνουμε το θέμα αυτό. Έκθεση της ε, κυρίας Τρίπελ για τον έλεγχο του Μητρώου των ε, ομάδων εμπειρογνώμων στην Κομισιόν Συμβαστική 1 που καλύπτει την τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 που καλύπτει την τροπολογία υπέρθυμο 2 της κυρίας Γκρέσλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 της συγκεκριάς υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία τε... Συμβαστική 3 που καλύπτει την 4 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία υπαριθμών 5. Ψηφίσατε όλοι πέρας πληροφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. 15-11. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Επτά. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση, λέει ο πρόεδρος. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται 15-15. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 9. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16-13. Τροπολογία 10. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4 που καλύπτει την τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 έχει αποσυρθεί. Έχει αποσυρθεί, λέει ο πρόεδρος. Δεν το εγνώριζε. Το σύνολο του κειμένου, λοιπόν. Με ονομαστική κλίση, παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ομόφωνα εγκρίνεται το κείμενο αυτό. Συγχαρητήρια στην κυρία Τρίπελ. Αγαπητοί μου συνάδελφοι, έχουμε εξαντλήσει την ημερησία διάταξη. Θα τα πούμε σήμερα το απόγευμα στις 3 για την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Διακοπή της συνεδρίασης.